Okay, colleagues, we're a little bit late. Συνάδελφοι, έχουμε αργήσει για αυτό το τελευταίο σημείο της μέσα διάταξης. Τελευταίο, αλλά σημαντικό είναι το υπαριθμό 17, η ολοκληρωμένη απάντηση, πλαίσιο και η εφαρμογή του για την Ουγγάντα. Είχαμε πάει κάποια από μέσα αποστολή στην Ουγγάντα. τα συζητήσαμε διαμακρών στην Επιτροπή. Επομένω, ε, έχει ε, σημασία και είναι επίκαιρο να συζητήσουμε αυτό το πλαίσιο της ολοκληρωμένης απάντησης προέκυψε κατόπιν συμφωνίας του 2016 κάποιες διακήρυξεις για πρόσφυγες και μετανάστες ε, σε συνεργασία με διάφορες πιλωτικές χώρες και κάποια από αυτές είναι η Ουγκάντα. Μπελίζε, Κωνσταντίζα Γουατεμάλα, Δούρα, Μεξικό, Παναμάς, Σομαλία, Τζιμπούτι, Αιθιοπία, Κένια, Ζάμπια, Ρουάντα και η Ουγγάντα. Οπότε η ουσία αυτή της ρύθμιση ε, πλαισίου, Πώ να το πούμε, ε, δράση θα το έλεγα εγώ, τελικά ο σκοπό είναι να υπάρχει επιτόπου ε, συντονισμό. Έχουμε ακούσει πολλέ ονομασίες, αλλά ένα σωρό φορεί εκεί, και φέρουν πόρους στις προσπάθειες, οπότε τελικά πρόκειται για κάποιο είδου απάντηση στο πρόβλημα που έχει, είναι συντονισμένη ε, και υποστηρίζουν όχι άμεσα τους ε, πρόσφυγες αλλά τις κοινότητες που τους υποδέχονται. Και διαπιστώσουμε ότι είναι 1,4 εκατομμύρια αυτοί οι οποίοι προσφεύγουν στην ε, Ουγγάντα. Πάρα πολύ από το Νότιο Σουδάν, συνήθως παιδιά και γυναίκες. Και να μην φιλιαρίσω άλλο, γιατί εδώ έχουμε τους ε, ειδικού μας, τον κύριο Μαμαντούνταν Μπάλτε, που είναι ο υποδιευθυντής της ε, αρμόδιας υπηρεσίας της υπάτης αρμοστίας για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ. Επίσης έχουμε την πρέσβυρα Μίριαμ Μπαξόου που είναι επικεφαλή αποστολή τη πρεσβείας τη Ουγγάντα ή στο Βέλγιο. Οπότε να δώσουμε το λόγο πρώτα στον, στον κύριο Μπάλντε και κατόπιν στην ε, ε, πρεσβεία και κατόπιν να ακούσουμε τους ε, συναδέλφους και επίσης να αναφέρουμε τα όσα μάθαμε στην αποστολή μας στην Ουγγάντα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να σας ε, παρουσιάσουμε το πώς στην πράξη εφαρμόζεται αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο, αυτή η απάντηση στο προσφυγικό, να, να δούμε τι πρόοδος έχει επιτευχθεί, τι προβλήματα έχουμε συναντήσει και να σας πω και εγώ πώς βλέπω το θέμα και θα συμπληρώσει και η κυρία Πρέσβης ε, που ευτυχώς είναι εδώ. Και πριν από 20 μήνες συμφωνήθηκε αυτό το πλαίσιο στην Νέα Υόρκη. Ήταν χωρίς προηγούμενο το πόσα κράτη, πόσοι αρχηγοί κρατών συμφώνησαν, ήταν 193 και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση των προσφύγων θα πρέπει να τους πλησιώσουμε όσο γίνεται καλύτερα, να τους δώσουμε κάποια ευκαιρία για αξιοπρεπή διαβίωση. 20 μήνες πέρασαν και είπα ότι η αρμοστία τώρα καλείται να εφαρμόσει αυτό το πλαίσιο, να υπάρξει κάποιο είδου ε, συνολικό παγκόσμιο σύμφωνο για να δούμε πώς μπορεί ο κόσμος μας να είναι πιο φιλικός προς ε, αυτούς τους ανθρώπους, τους ε, πρόσφυγες. Οπότε ευθύς εξ αρχής να σας πω δύο λόγια. Περί τίνος πρόκειται. Τι είναι αυτό το πλαίσιο. Έχει τέσσερες στόχους που θα πρέπει να επιδιώξουμε ε, που να προσπαθήσουμε για όλους. Για κάποιες χώρε όπω η Αιθιοπία, η Λίβων, η Αιθιοπία, η Ιορδανία, για αυτέ τι χώρε θα πρέπει να τι ανακουφίσουμε από την πίεση που υφίστανται λόγω του μεγάλου ρυθμού των προσφύγων και έχουμε πολλά μέσα προς το δεύτερο στόχο, ότι αφού τις ανακουφίσουμε από την πίεση που υφίστανται θα πρέπει να είναι οι πρόσφυγες κάπως πιο αυτόνομοι για να μπορέσουν να ζήσουν ε, και να συμβιώσουν με αυτούς που τους φιλόξενουν μια ε, ε, κάποιο είδους ε, αξιοπρέπεια. Τρίτος στόχος είναι να ε, υπάρχει κάποια μετεγκατάσταση και τότε είναι κάτι να κάνουμε με τις χώρες της προέλευσης, να δημιουργήσουμε συνθήκες για να μπορούν να γυρίσουν οι πρόσφυγες. Αυτά όσον αφορά αυτό το πλαίσιο και όλοι υποσχεθήκαμε ότι θα το υλοποιήσουμε και το συμφωνήσαμε το Σεπτέμβριο του 2016. Οπότε κάνουμε αυτή την διαδρομή αυτή την προσπάθεια του τελευταίους 20 μήνες. Συνεργαστήκαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε διάφορες αντιπροσωπείες ε, σε διάφορα επίπεδα και περιφερειακά επιληφθήκαμε και οπότε υπήρξε ανθρωπιστική υποστήριξη, αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά να σταθούμε λίγο περισσότερο στο τι ανάγκες συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν πιστώνω ότι και εσείς τα βλέπετε με τα μάτια σας γιατί πήγατε στην ε, Ουγκάντα. Οπότε ε, πρέπει πραγματικά να διαπιστώσουμε ότι συνεργαζόμαστε για αυτό το σκοπό. Μετά τη διακήρυξη λοιπόν της Νέας Υόρκης υπάρχουν κάποιες πάρα πολύ καλές πρακτικές. Πρώτα-πρώτα να εφαρμόζουμε σε περιφερειακό επίπεδο αυτό το πλαίσιο, όπως το Ανατολικό κύριο της Αφρικής και εκεί να συνδυάζουμε τις προσπάθειες για Κένια, Ουγγάντα, Αιθιοπία, Τζιμπουτή και για κάποιες άλλες χώρες. Και έτσι να είναι κοινή η προσπάθεια για να κάνουμε κάτι στο μέτωπο της ε, Σομαλίας και να έχουμε τον επαναπατρισμό, τον εθελοντισμό, να φέρουμε τις χώρες να βοηθούν τους πρόσφυγες να μπορούν να έχουν γη, νερό, αξιοπρέπεια, ε, ελεύθερη διακίνηση και η κτήθης εμπειρία ήταν πάρα πολύ ε, αξιόλογη. Μεξικό, Κεντρική Αμερική και εκεί είχαμε χώρες ε, ασύλου διαμετακόμισης, προέλευσης, οπότε προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε πρόσφυγες να καλυφθούν. Κάποιοι ρώτησαν για τις επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις που διαπιστώνουμε είναι πολλές. Κάποιες έχουν να κάνουν με αλλαγή της πολιτικής. Γιατί κάποιες χώρες όπως το Τζιμπουτί άλλαξαν τελείως την πολιτική τους και σήμερα επιτρέπουν την εργασία στους πρόσφυγες και την ελεύθερη διακίνησή τους. Άλλαξαν το δίκαιό τους και έχουν θεσπίσει κάποιους ε, νόμους τους οποίους εφαρμόζουν. Και οπότε υπάρχει αυτή η επιπλέον ε, βοήθεια, αλλά και στην ε, Ουγγάντα. Εκεί έχουμε 40 εκατομμύρια και πρόσφυγες γύρω στο 1,4 εκατομμύρια. Και εκεί συνεχίζεται αυτή η πολιτική υποστήριξη και οπότε αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά ορόσημα, αυτά που πετύχαμε, γιατί συνεχίζονται οι ζωές των προσφύγων. Α, πρόκειται περί κάποιων θετικών προσπαθειών και πολιτικών. Στη Κωνσταντίνα οι πρόσφυγες επίσης ε, ε, δέχονται βοήθεια όπως και ο τοπικός πληθυσμός για να αντιμετωπίσουν την φτώχεια που τους μαστίζει και τέλος και εδώ θα βάλω τελεία σε αυτό το τμήμα είναι το τι προσπάθειες γίνονται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Δύο δις για τους αμφιτρίωνες αλλά και για τους ε, πρόσφυγες. Η ΔΕΦΚΟ προσπαθεί και υπάρχουν συγκεκριμένοι ε, μηχανισμοί που θέλουμε να συνεχιστούν και να αναβαθμιστούν και διμερός έχουμε από Νορβηγία και άλλες χώρες να υπάρχει υποστήριξη. Αυτά όσον αφορά την επιδεχθήσα πρόοδο. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Θα σας τα πει και κύριε Πρέσβες, αλλά παιδεία και υγεία σε κάποιες χώρες όπως η Ουγγάντα ε, είναι τομεί που ε, υπάρχουν ανάγκες. Αυτό αφορά για το, νερό, χρειάζεται ανθρωπιστική αρρωγή, Πάντω ενώ περιμένουμε ε, τους καρπούς της ανάπτυξη θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τη βοήθεια να είναι προσπάθεια βιώσιμη, να βοηθήσουμε επομένως για παιδεία, για νερό, υποδομές πολλές φορές. Ε, υπάρχει ανάγκη οποία συνεχίζει να υφίσταται τώρα όσον αφορά τις πολιτικές διεργασίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να σταματήσουν οι ζωές των προσφύγων ή να μειωθούν. Εκεί δεν υπάρχουν τόσα κεφάλαια. Ε, υπάρχει κάποια πρόοδος, να συνεχίζουν να έρχονται οι πρόσφυγες και από τις χώρες προέλευσης συνεχίζεται η ροή των προσφύγων και πηγαίνουν στις όμορες χώρες όπως η Ουγκάντα όπου δεν έχουμε δημιουργία συνθήκων για αυτές τις αυξανόμενες ροές. Για να ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη εισήγηση, να σας πω ότι αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο απάντησης είναι μία από τις καλύτερες ευκαιρίες που είχαμε για να παρεύουμε στο προσφυγικό. Πολλές χώρες έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Και η Ουγγάντα. Αλλά έχουμε την αύξηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά συνεχίζει και χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια. Γι' αυτό και η, η του ΟΗΕ δεν θα σταματήσει αυτή τη διαδρομή, αυτή την ε, προσπάθεια. Αυτά από μένα και φυσικά ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε. Η κυρία Πρέσβης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε σήμερα και στη συζήτηση αυτή για την κατάσταση των προσφύγων με κύριο αντικείμενο την Ουγγάντα Θα γνωρίζουν πολλοί από εσά ότι μέχρι μερικές δεκαετίες πριν η Ουγγάντα ήταν η ίδια πηγή προσφύγων με χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδων προσφύγων εκτός της Ουγγάντα κατά, την, ε, κατά το καθεστώς του Ιντία Μινταντά και βεβαίως στη συνέχεια και υπό τον πρόεδρο Μουσέβενη ο οποίος μπήκε στην Ουγγάντα το 86. Τώρα ευτυχώς είναι σταθερή χώρα. Η Ουγγάντα. Όσοι έχουν εμπειρία από την προσφυγιά, έχοντας ζήσει έξω από την Ουγγάντα, ξέρουν ότι δεν πρέπει ποτέ να ξαναζήσει κανείς. Ε, δεν πρέπει να ε, ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Επομένως στηρίζουν τις γειτονικέ χώρες. Η κυβέρνησή μου είναι προσιλωμένη να συνεχίσει να προστατεύει εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σε άλλες χώρες και τους καλωσορίζει. Αυτό απαιτεί βεβαίως και την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ουγγάντας. Ε, εγχείρημα όχι ευχερές, διότι καλούμε τις ε, τοπικές κοινότητες να προσφέρουν γη ώστε να εγκατασταθούν εκεί οι πρόσφυγες. Ή σε ένα πρώτο στάδιο ζητούμε να τους προσφερθεί νερό, τα είδη πρώτης ανάγκης. Και μέχρι στιγμή αυτό έχει φέρει αποτελέσματα. Βεβαίω έχουμε περάσει από ένα πληθυσμό των 400.000 σε 1,4 και άνω εκατομμύρια μέσα σε ένα μισή χρόνο, και αυτό σημαίνει τεράστια προσπάθεια, όχι μόνο για την κυβέρνηση Ουγκάντας, αλλά και για τους αναπτυξιακούς μας εταίρους, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπή χορηγή. Ενισχυμένη λοιπόν η υποστήριξη είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Δεν χρειάζεται νομίζω να εξηγήσω περισσότερο την, ε, το συνολικό πλαίσιο ανταπόκριση στο προσφυγικό, όπως εξήγησε ο κύριος ε, Ντεμπάλτε, με τους τέσσερις πυλώνες. Είμαστε απολύτως προσιλωμένοι σε αυτό. Αλλά χωρίς υποστήριξη και μια, έναν πιο ισότιμο επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ της Ουκάνδας και της Εθνούς Κοινότητας δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Έχουμε εγκαταστάσεις, δεν τις ονομάζουμε καταφλισμούς. Πιστεύω έχετε αντιληφθεί τη διαφορά. Τους προσφέρουμε νερό, τροφή, ε, αρμοστία, πρώτα, πρώτες ύλες και υλικά για να το χτίσουν μόνοι στα σπίτια τους. Ωστόσο, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα μπροστά μας, την κλιματική αλλαγή, η οποία έχει αλλάξει πολύ το οποίο είχαμε τις τελευταίες έξι εβδομάδες νερό, όσο δεν είχαμε δει ε, για πολύ καιρό. Μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε πολλές ε, κατολιστήσεις. Δεν συνέβη αυτή τη φορά, αλλά χάνουν ε, γη γενικά οι πολίτες και αν δεν χάσουν γη χάνουν, καταστρέφεται η παραγωγή τους ή τα σπίτια τους. Ό,τι έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν και στο βορρά όπου είδαμε απότομες βροχοπτώσεις, τα στατιάς που κατέστρεψε τη συγκομιδή, ευθύνουν τώρα και αυτοί έτοιμο προς ε, βοήθεια, για βοήθεια προς την κυβέρνηση. Επομένως, ναι, έχει μάθει η Ουγκάντα και υποδέχεται τους πρόσφυγες, αλλά όταν και ο ντόπιο ε, χωρίς πληθυσμός αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα, μένει χωρίς δουλειά, μένει χωρίς σπίτι, μένει χωρίς τα προστοζήνα ή πόρους, ε, ακόμα και αν δεν είναι εξόριστος ή αν δεν έχει εκδιωχθεί από το σπίτι του, δεν έχει σπίτι, ναι, άρα στις ίδιες συνθήκες με τον πρόσφυγα. Και αυτό σας το λέω για να δείτε και την εικόνα, φανταστείτε τώρα μια μεγάλη ε, αυτοκινητοπομπή φορτηγών της ΥΠΑ της αρμοστίας που πηγαίνει στις εγκαταστάσεις που έχουμε για τους πρόσφυγες με όλα τα απαραίτητα τρόφιμα, νερό και τα λοιπά και περνάει μπροστά από του Ουγγαντέ αυτού που έχουν χάσει τα σπίτια του και αυτοί λένε Μα και εμεί χάσαμε τα σπίτια μα, γιατί δεν έχουμε εμεί τέτοια περιποίηση, γιατί πάνε μόνο στου άλλου. Και κάνω απεγνωσμένε προσπάθειε σε σχέση και με του υπουργού και των οικονομικών και του λοιπού να ζητήσω επιπλέον χρηματοδότηση για να ε, προσφερθεί η υποστήριξη που χρειάζονται οι ε, Ουγγαντινοί. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια, αλλά όπως είπα και ναι μεν είναι θετικό το κλίμα έναντι των προσφύγων, αλλά οι αλλαγές, οι κλιματικές, μπορούν να φέρουν και άλλες αλλαγές. Και εδώ θέλω να σταθώ στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, να τηρηθούν οι στόχοι για την κλιματική αλλαγή. Ε, είχα πέρσι ε, την πληροφορία σε μια επίσκεψή μου εκεί ότι μια οικογένεια προσφύγων χρειάζεται μισό δέντρο την ημέρα. Δηλαδή, ε, μέρα την ημέρα πρέπει να κόβεται από μισό δέντρο για κάθε οικογένεια για να εξασφαλιστούν οι ανάγκε τη ε, σε, σε ξύλα, καυσόξυλα, για τα, η ντροφή της κτλ. Λοιπόν, ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε σε συνεργασία με διάφορους φορείς να βρούμε πιστώσεις, άνθρακα, ώστε να μην χρειάζεται να κόβουν τα δικά μας δέντρα ή να κόβουν τις, ε, το ψηλό χόρτο που χρησιμοποιούμε για να φτιάχνουμε σπίτια, γιατί αυτές οι καλύβες είναι φτιαγμένες με, χόρτο. και βεβαίως αυτό είναι κατεπήγον να γίνει πριν χαθούν όλα τα δάση της Ουγκάντας από το βορρά τουλάχιστον. Ε, ο κύριος Ντεμπάλτε μίλησε για την εκπαίδευση ε, και εγώ την επισκέφθηκα την περιοχή. 100 παιδιά μέσα σε μία τάξη, ούτε θέση να κάτσουν δεν έχουν, ούτε καν στο πάτωμα ε, δεν έχουν χώρο να κάτσουν. Γίνεται πρωινό και απογευματινό σχολείο. Πολλές οικογένειες ζουν χωρίς πατέρα η σύζυγο και έτσι έχουν γίνει πια αρχηγοί της οικογένειας οι μητέρες, οι σύζυγοι, οι γυναίκες και άρα πρέπει να σταθούμε και σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να μπορούν και οι γυναίκες αυτές να σταθούν στα πόδια τους, να κάνουν μια δουλειά, να κερδίσουν τα προστοζήν για τις οικογένειές τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, πέραν βέβαια και της κοινωνικο-ψυχολογικής υποστήριξης. Ε, θεωρούμε βέβαια, ξέρετε, στην Αφρική ότι ο καθένας έχει να ξεπεράσει μόνο στα ψυχολογικά του προβλήματα, αλλά πάλι είναι άνθρωποι όσο και οι Ευρωπαίοι δηλαδή, μας, ε, είμαστε άνθρωποι όσο και οι Ευρωπαίοι, άρα μας τραυματίζουν ε, ψυχικά οι εμπειρίες μας όσο και τους Ευρωπαίους. Αν δει κάνει μια γυναίκα τον άντρα του να δολοφονείται, εάν έχει χρειαστεί να φύγει από τον Νότιο Σουδάν διωγμένη, αν έχει δει την κόρη της να βιάζεται, προφανώς έχει τα ίδια προβλήματα και το, το ψυχικό τραύμα και το άγχος ε, που μεταφέρει μαζί της και βλέπω ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη κοινωνικο-ψυχολογική υποστήριξη αυτή τη στιγμή. Ε, δεν ξέρω αν έχω ξεπεράσει τα χρονικά όρια που μου έχετε διαθέσει. Είναι πολλές ε, οι προκλήσεις, σας τις αναφέρω και χωρίς τη δική σας υποστήριξη δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα για τους ε, πρόσφυγες που υποδεχόμαστε το τελευταίο 1,5 χρόνο με τους όρους που έχουμε μπορέσει μέχρι τώρα να τους εξασφαλίσουμε. Βέβαια συνεχίζουμε τις επαφές με τους εταίρους. Είμαστε ένα σύννεφο σταθερότητα θα έλεγα, στην περιοχή. Αλλά έχουμε μεγάλα προβλήματα. Έχουμε και την γειτονική λαϊκή δημοκρατία του Κόγκο. Έχουμε πρόσφυγες που καθημερινά φτάνουν. Έχουμε πρόσφυγες από τον Μπουρούντι. Σήμερα γίνεται δημοψήφισμα στο Μπουρούντι και δεν ξέρουμε τι θα προκύψει από εκεί. Πάντως η κατάσταση γύρω μας, στις γειτονικές χώρες, δεν είναι σταθερή και έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο Νοτιοσουδανού που όμω εξακολουθούν να έρχονται διασχοντίζοντα τα σύνορα γιατί δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση του Νότιου Ο πρόεδρο μου, η κυβέρνησή μα κάνουν μεγάλε προσπάθειε ώστε να ε, ζητούν, να επιδιώκουν, να υποστηρίζουν διαρκώ ειρηνικέ λύσει σε σχέση με τι χώρε που μα ε, περιβάλλουν δεν έχουν ακόμη επιτύχει. Απευθύνουμε έκκληση λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά τη διεθνή κοινότητα να μας τρίχουν στην προσπάθεια για την επίτευξη ειρηνικών λύσεων στις χώρες εκείνες από τι οποίε προέρχονται οι πρόσφυγες. Και οπωσδήποτε αυτό διότι μόνο μία βιώσιμη και διαρκή, ε, ότι μία βιώσιμη και λύση ε, μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με την εθελοντική επάνωδο, τον εθελοντικό επαναπατρισμό των προσφύγων αυτών και στέκομαι σε αυτό, επιμένω σε αυτό, γιατί θα επαναπατριστούν εθελοντικά οι άνθρωποι αυτοί μόνο όταν έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες της χώρας τους. Ευχαριστώ πολύ. Είδαμε πολλά από αυτά που μόλις περιγράψατε, για παράδειγμα το πρόβλημα ε, του διαμερισμού του ξύλου, της τοπικής ξυλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει σε συνεργασία με ε, ΜΚΟ ε, στην χρήση ειδικών πετρών για, την, για, την, για να μαγειρεύουν οι ντόπιοι πληθυσμοί γιατί θα υπάρξει πρόβλημα έλλειψης ξυλίας και κύριε ε, Πρέσβερα είπατε ότι ε, αυτοί που ζητάμε από αυτούς που έχουν λίγα να μοιραστούν ε, τα λίγα που έχουν με αυτούς που δεν έχουν τίποτα. Και είδαμε παιδιά με πολύ μεγάλο ψυχικό τραύμα, κορίτσια 12-13 ετών. Στην αρχή δεν μιλούσαν και μετά ε, άρχισαν να εκφράζονται. Πρόκειται για έφηβες που έχασαν τους γονείς τους, που ε, είδαν ε, σκηνές ομής βίας, είναι ευάλωτες νεαρές γυναίκες. Και με τους υπουργούς με τους οποίους συζητήσαμε ήταν, υπήρξαν οι ίδιοι πρόσφυγες ε, είχαν, ε, πολλοί από αυτούς είχαν πάει στο Σουδάν, οπότε κατανοούσαν ε, τη κατάσταση στην Ουγγάντα Μιλήσαμε ανοιχτά για τα προβλήματα που εντοπίζουν οι ντόπιοι πληθυσμοί. επειδή στο Νότιο Σουδάν υπάρχουν πολλά προβλήματα, εισραίουν οι μετανάστες και υπάρχει πρόβλημα δημόσιας υγείας. Πολλά παιδιά που έρχονται δεν έχουν εμβολιαστεί. Την πόλη μου βλέπω ε, άτομα, ανθρώπους να έρχονται και έρχονται, ε, φέρνουν ασθένειες. Υπάρχει πρόβλημα με το εκπαιδευτικό σύστημα. Κάποιος από του υπουργού είπε ότι ένας δάσκαλος του είχε πει ότι ουσιαστικά το να διδάσκει είναι σαν να ελέγχει απλώς ένα πλήθος ε, παιδιών. Υπάρχουν τεράστιε ανάγκες λοιπόν στο τομέα τη εκπαίδευση. Είχαμε την εντύπωση ότι αυτό το πλαίσιο ολοκληρωμένης απάντησης είναι το κατάλληλο για την ε, πρόθεση της συμβίωσης των τόπιων πληθυσμών με τους ε, πρόσφυγες βλέπουν και οι ντόπιοι πληθυσμοί πώς μπορούν να υποφεληθούν από αυτό το πλαίσιο ολοκληρωμένη απάντηση και στην Μέση Ανατολή και στο Λίβανο παρατηρούμε εντάσεις γιατί πρόσφυγες λαμβάνουν κουπόνια και έχουν παραπάνω να ε, δαπανίσουν από τους ντόπιου πληθυσμούς και στην Ελλάδα ε, Υπάρχουν τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και κάποιοι βλέπουν ε, πρόσφυγες να λαμβάνουν στέγη ε, χωρίς, ε, χωρίς να ξοδεύουν τίποτα και είναι απαραίτητο να δοθεί μια απάντηση από πλευράς του ΟΗΕ σε αυτό το πρόβλημα Το ίδιο όμως δεν ισχύει με τις κοινότητες προσφύγων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. θα βοηθούσε να χρηματοδοτηθούν δράσεις και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις που παρατηρούνται απέναντι στους πολιτισμούς προσφύγων. προσφύγων. Σε κάποιες χώρες πάντως υπάρχουν πολύ μεγάλοι αριθμοί προσφύγων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει η απαραίτητη κατανομή των ε, πληθυσμών προσφύγων. Ε, στη Έχει το λόγο για να κάνετε τις, ε, τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ Λίντα, ευχαριστώ πολύ τους σημερινούς μας καλεσμένους πολύ ε, ενδιαφέρουσα εμπειρία η αποστολή στην Ουγγάντα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας κάτι που αναφέρουμε πολλές φορές ε, στην Ουγκάντα. Υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στην Ουγκάντα και η χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μόνη της. Και είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγα ότι έχει αιμονή πραγματικά με τις ροές μεταναστών από την Αφρική ιδιαίτερα. Έχω την εντύπωση ότι στα πλαίσια αυτής της συζήτησης ξεχνάμε ότι η πλειοψηφία των εκτοπισμένων ατόμων ε, φιλοξενούνται από ε, ε, χώρες. Πρέπει να το λόβουμε υπόψη μας. Ε, ήμουνα και εγώ στη Νέα Υόρκη ε, στην ε, Σύνοδο. Η καλύτερη υποδοχή των προσφύγων είναι παγκόσμια πρόκληση. Δεν πρέπει να την αντιμετωπίσει μόνο η Ευρώπη και έχουμε ευθύνες. Αυτό που είδαμε είναι μια πολύ προοδευτική πολιτική που βλέπει τη χορήγηση γη στους πρόσφυγες και για να παραθέσω κάτι που είπε ένας από τους ηγέτες, ήμασταν κάπου στο Αλέρε και ο ο αρχηγός της ε, ε, κοινότητας προσφύγων και της, ε, το, των ντόπιων μα, μιλούσαν μαζί μας και ο, ο αρχηγός της ντόπιας κοινότητας είπε ότι υποδεχόμαστε τους αδερφούς μας. Ε, ε, έχουμε, γνωρίζουμε το παρελθόν μας και δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας ε, περιμένει, τι μέλη γενέστε. Άρα μοιραζόμαστε το μέλλον μας με τους, αδερμό, αδερφούς μας προκειμένου να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς και να μην είναι σαν ζητιάνοι. Είναι πολύ σημαντικό μήνυμα αλληλεγγύης ανάμεσα στον ντόπια, πληθυσμό και την κοινότητα των προσφύγων επισκεφτήκαμε επιτόπου διάφορες εγκαταστάσεις όπου υλοποιούνται δράσεις στις οποίες συμμετέχουν και ο ντόπιο πληθυσμός και οι πρόσφυγες. Εκεί όλοι οι φορείς καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να ανταποκριθούν στις ε, ανάγκες σε συνεργασία με τους, με και με την κυβέρνηση όπως ε, είπατε στα πλαίσια ενός εθνικού σχεδίου δράσεως. Γνωρίζουμε ότι αυτό το σχέδιο δράσης λαμβάνει υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, πολύ καλό αυτό, και ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αυτή τη στιγμή, πρέπει να ε, ε, συμμετέχουν περισσότερο και άλλες ε, χώρες. Είναι απαραίτητο αυτό. Οι εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο είναι ανασυχητικές. Η κρίση μπορεί να επιδεινωθεί και η Ουγγάντα έχει φτάσει τα όρια της. Πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες. Πρέπει να προσφέρουμε μεγαλύτερη υποστήριξη σε τρεις τομείς. Την υγεία, θα έλεγα πρώτα απ' όλα, γιατί επισκεφτήκαμε κέντρα υγείας που είναι εξαιρετικά στην Ουγγάντα και παρά τις προσπάθειες ε, που υποδέχονται 200 άτομα ε, την ημέρα είναι πολύ απομακρυσμένο. Είναι δύσκολο να χορηγηθεί ε, ιατρικό, φαρμακευτική περίθαλψη και στις εγκαταστάσεις των προσφύγων και στο τομέα της εκπαίδευσης επισκεφτήκαμε κάποια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 200 παιδιά 100 παιδιά για έναν δάσκαλο κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολες τέτοιες συνθήκες για να ε, ε, δοθεί απαραίτητη εκπαίδευση. Χρειάζονται περισσότερες εγκαταστάσεις, περισσότεροι δάσκαλοι και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί όλοι οι φορείς επιτόπου μας είπαν ότι υπάρχει και εκεί μεγάλο πρόβλημα και δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Και κάτι ακόμα, τα τρόφιμα. Γνωρίζουμε ότι το Παγκόσμιο Επιστημιστικό ε, Πρόγραμμα αντιμετωπίζει προβλήματα, μπορεί να χρειαστεί να ε, μειώσει την υποστήριξή του, κάτι το οποίο θα ήταν καταστροφικό. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες και σε αυτό το τομέα, γιατί Όποιες και αν είναι οι δυσκολίες πρέπει να φροντίσουμε να ε, μειώσουμε τις ε, κοινωνικές εντάσεις ό,τι αφορά την ε, παροχή τροφίμων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Θα είναι χαρά μας να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και τις συζητήσεις μας και κάτι ακόμα να τονίσω σε αστικό περιβάλλον έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχουν λιγότερες ανησυχίες ή τουλάχιστον δίνονται λιγότερες απαντήσεις για να, ε, να δοθούν απαντήσεις ανάγκες προσφύγων που έχουν μετακινηθεί από τις εγκαταστάσεις σε αστικά κέντρα. Είναι απαραίτητο να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν Α, έχει ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Τσέλερ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Όντως, Πρέπει να βοηθούμε τους πρόσφυγες και στην επιβίωση, αλλά και βεβαίως να τους υποδεχόμαστε στα κράτη. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και ποια είναι η ρίζα της προσφυγέας. Γιατί ο Σαλβακίρ και ο Ρίκ Ματζάρ δεν πλήττονται από κυρώσεις, γιατί τους αφήνουμε, γιατί έχουν πλουτίσει από τον πόλεμο. Αγοράζουν πολυτελείς επαύλη στο εξωτερικό, γύρω από το, στην πιο ακριβή γειτονιά του Ναϊρόμπι, το πιο ακριβό προάστιο, έχουν βίλες και δεν ε, τους πλήττει κανείς. Ενώ για άλλους είμαστε έτοιμοι να επιβάλλουμε κυρώσεις. Όταν είναι σαφές ότι είναι ε, έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην περίπτωση όμως αυτοί δεν κάνουμε τίποτα και ίσως άμα φύγουν αυτοί από τη μέση να σταματήσουν και τα δεινά των πολιτών. Είναι διπλό το καθήκον μας λοιπόν. Να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες, τα κράτη που τους υποδέχονται, αλλά πρέπει σιγά σιγά και να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση εναντίον εκείνων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα δεινά των ανθρώπων αυτών. Αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να κόψουμε τη ροή του παράνομου ή και του νόμου χρήματος που φτάνει στα χέρια τους, αν δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αποξήρανση του σιπήριν αυτής της, ε, ε, αυτού του πακτολού, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Yeah, I mean very clear that the conflict in South Sudan. Είναι σαφές το ότι η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν, αυτός είναι φίλος πόλεμος, θα πρέπει να λάβει τέλος, γιατί ακριβώς ανθίζει το λαθρεμπόριο όπλων και ανέκαθεν υπήρχαν εκεί αυτές οι αντιμαχόμενες πλευρές και χρειάζεται κάποια πολιτική λύση στην περιοχή και στη ζήτηση με τον Επίτροπο το τονίσαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει σφαιρική αντιμετώπιση τι γίνεται στο Κονγκό, τι γίνεται στο Μπουρούντι χτες συζητήσαμε για το Σουδάν, στο Νότιο Σουδάν, ένα ε, χρεοκοπημένο κράτος και την Ουγγάντα σχεδόν σε αυτό, το επιβάλλεται η πολιτική λύση. Καθώς μάλλον είχα και την ευκαιρία να παρακολουθήσω ως παρατηρητής ε, το δημοψήφισμα που δείξε σε ανεξαρτησία στο Νότιο Σουδάν και είδα η ε, μας τον ενθουσιασμό των ανθρώπων θεώρησαν ότι με το δημοψήφισμα αυτό και την αυτονομία εξασφάλιζαν την ε, απαλλαγή τους από τη δουλεία και δεν έγινε τίποτα. Κάποιοι μάλιστα έχουν φτάσει να λένε ότι μπορεί η αναγνώριση ανεξαρτησία για τον Νότιο Σουδάν να ήταν λάθος και ότι πρέπει ίσως να επανενωθεί με το Βόρειο Σουδάν. Και αυτό ασφαλώς θα ήταν τεράστιο σφάλμα, έχοντας υπόψη βέβαια τι είδους καθεστώ επικρατεί στο Βόρειο Σουδάν. Είπα το μαγικό ραβδάκι. Μακάρι να ήταν έτσι και έτσι όλα να ρυθμιζόντουσαν. Τόσα χρόνια υπάρχει αυτό το πρόβλημα στο Νότιο Σουδάν και μετά την ανεξαρτησία αναδείτε, ξαναναδείτε το πρόβλημα. τέλο πάντων, ε, τι έχετε να πείτε. Κύριος, είσαι εσείς κυρία Πρέσβη για τι ερωτήσει. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ του βουλευτέ που έλαβαν τον ε, λόγο για να δεις τι παρατηρήσεις τους και νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο μικρό σχήματος για το πώς έχει η κατάσταση και για το τι επιβάλλεται να γίνει αλλά είναι θέμα χρημάτων αναζήτηση λύσεων για τις πολιτικές συγκρούσεις στις γειτονικές μας χώρες αλλά αυτό προβληματίζει πάρα πολύ τον πρόεδρο. Επιδεινώνει την κατάσταση του Νότιου Σουδάν και σήμερα κυβερνά όποιος έχει το όπλο στο χέρι. Τόσο πολλές ενημαχωμένες μερίδες υπάρχουν εκεί. Και βλέπουμε η σύγκρουση να πάρω ξύντε να χειροτερεύει απέσια κατάσταση και όπως είπε η κυβέρνηση είπαμε όχι σε εμπάργο και σε κυρώσεις τώρα όμως ε, κάναμε στροφή τώρα λέμε ναι σε τέτοιες κυρώσεις να υπάρξει έλεγχος των όπλων γιατί κυκλοφορούν περισσότερα όπλα και έτσι επιδεινώνεται η κατάσταση άρα διεθνής πίεση, εμπάργο, κυρώσεις. Οπότε έτσι τουλάχιστον να μην χειροτερεύουν τα πράγματα, τουλάχιστον να μην η κατάσταση όπως έχει και να ψάξουμε για κάποια λύση. Να δούμε τι θα γίνει στο κέντρο της Αφρικής, τι θα γίνει στο Νότιο Σουδάν και κατά τον εμφύλιο του Σουδάν είχαμε 200-300 χιλιάδες ε, πρόσφυγες που έμειναν μια δεκαετία και πάνω. Και μετά την εξαρτησία του Νοτιού Σουδάν νιώσαμε μεγάλη ανακούφιση που επέστρεψαν. Όμως η σημερινή κατάσταση τους οδηγεί να ξαναφεύγουν από τη χώρα. Είναι ένα κράτος εν διαλύσει, άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Και επίσης το ίδιο προβληματικό είναι και το Κονγκό. Είναι τόσες ε, οι αντιμαχόμενες ομάδες εκεί και πολλές φορές έχουμε αυτή την στη διεθνή κοινότητα και υπάρχει και κάποια ομάδα ADF ε, Allied Defense Forces που κάνει επιδρομές κατά της ε, Ουγγάντα. νομίζαμε ότι βρίσκονται υπό έλεγχο είναι φονταμεταλιστές, Ισλαμιστές πολύ επικίνδυνοι Οπότε και εκεί όλοι αυτοί οι ένοπλοι διώχνουν τον κόσμο. Αναγκάζει τον κόσμο να φύγει, τους λαιλατούν. Πολύ θλιβερή κατάσταση. Όμως δεν θα σταματήσουμε τις προσπαθίες μας. Δεν θα σταματήσουμε να ζητούμε λύσεις. Και στο Μπουρούντι θα πρέπει να μπει μια τροχοπέδη στο θέμα. Επέστρεψαν ή αν τέλο πάντων επιστρέψουν όλοι αυτοί από τον Μπουρούντι που έχουμε θα είναι για μέσα ανακούφιση. Πάντως είναι η κατάσταση πολύ ευάλωτη, πολύ δύσκολη πολιτικά. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει υποστήριξη έως ότου σταματήσουν οι σύγκρουσεις. Μας πιέζει ο χρόνος, λέει. Ναι, να σας πω. Δύο λόγια και εγώ ευχαριστώντας σας πολύ σύντομα καταρχάς. Αν κοιτάξετε τον Νότιο Σουδάν, μετά το 72, από το 56 μέχρι το 72 είχαμε μεγάλο ρεύμα προσφύγων που επαναπατρίστηκαν όταν η κατάσταση βελτιώθηκε μέχρι που ξανά επιδεινώθηκε. Αυτό που αναφέρετε εσείς βεβαίως είναι όχι ανθρωπιστική αλλά πολιτική λύση. Εσείς έχετε ρόλο να διαδραματίσετε, να λάβετε τις αποφάσεις αυτές, τις πολιτικές σας, οι βουλευτές, στηριζόμαστε στη δική σας και περιμένουμε τις δικές σας επιλογές. Ε, κλείνοντας μόνο, δεν θέλω να πω τα εξή. η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν είναι στο 6% και από ό,τι μας λέει η Πατιαρμοστή έχουμε ένα 9% μόνο ε, παναπατρισμού ή αποκατάσταση. Ε, έτσι λοιπόν ακόμα και να σταματήσει τώρα η κρίση πάλι θα χρειαστεί η υποστήριξη για την επανεγκατάστασή τους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα στις κοινότητες που τους υποδέχονται. Η Πρόεδρος θέλει να πει κάτι. Ναι, βεβαίω. Είχαμε την Σύνοδο Αλληλεγγύη στην Ουγγάντα πέρσι και ασφαλώ θα γνωρίζετε κι εσεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια οργάνωση η οποία έδωσε υπόσχεση για 96,7 αν δεν απατώμε δισεκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίω αισθανθήκαμε μεγάλη χαρά για τη δέσμευση αυτή για την υπόσχεση αυτή, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώ που, πώς ε, επιμερίστηκαν τα χρήματα. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Ναι, δυστυχώς. Ωστόσο, περάσανε μέσα από, τις, ε, από τους φορείς, είπατε, αρμοστία και άλλους, τα κονδύλια αυτά. Εγώ από τη δουλειά μου εδώ στις Βρυξέλλες ξέρω ότι το καταπήγον καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική ε, θεσπίστηκε και είχαμε αμέσως ε, και στην αρχική ε, φάση 29 εκατομμύρια για, τον νότιο, για τους νότιους Σουδανέζους και μετά ακόμα 10 εκατομμύρια. 1,9 δις ευρώ έχει αυτό το καταπίστευμα. Ε, είναι τεράστιο ταμείο δηλαδή και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να αποδεσμεύει κονδύλια από το συγκεκριμένο αυτό ταμείο Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει περισσότερο τους Σουδανούς. Εδώ είναι η Κομισιόν. Δεν ξέρω αν μπορώ να του απευθύνω σήμερα το ερώτημα. Η κυρία Κόλλιο και ο κύριος Τρεβίσαν από την Τεύκο. Αλλά δεν έχω και πολύ χρόνο. Πάντως αν μπορείτε να δώσετε μια απάντηση και σας ευχαριστώ που μας βοηθήσατε στην προετοιμασία αυτής της αποστολής. Ήταν εξαιρετική η δουλειά σας. Μας βοήθησε πολύ. Ποιο θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ σύντομα. Ναι, πολύ σύντομα σε ό,τι αφορά τη, ε, δέσμευση για την υποστήριξη των ε, προσφύγων και των ντόπιων ε, πληθυσμών. 20 εκατομμύρια ήταν το αρχικό ποσό για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την ε, βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, τη τελευταία λειτουργική επιτροπή ε, του καταπεστηματικού ταμείου ε, με επιπλέον 20 εκατομμύρια για την υποστήριξη δράσεων σε συνεργασία με την γερμανική κυβέρνηση που δεσμεύτηκε να χορηγήσει 10 εκατομμύρια και δράσεις ε, στην Καμπάλα και στην περιοχή της Καμπάλα, όπου, ε, οι οποίες υποδέχονται ε, μεγάλους αριθμούς προσφύγων. Και θα έλεγα ότι σχετικά με όσα είπατε για την ανάγκη να υποστηρίξουμε και τους ντόπιου πληθυσμού και τις, τους πρόσφυγες, θα ήθελα να σας πω ότι στα πλαίσια των εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων και όλων των δράσεων πάντα στοχεύουμε αυτές τις δύο ομάδες πληθυσμού και στην Ουγγάντα ε, τρέχουμε ένα ακό πρόβλημα, ε, πρόγραμμα ε, επιστημιστική ασφάλεια μεταξύ άλλων ε, προκειμένου να ενισχύσουμε τη δράση της ε, κυβέρνησης για μας είναι πολύ σημαντικό και για την μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. Πάντα στόχος μας είναι υποστήριξη των ντόπιων πληθυσμών και των προσφύγων και δρομολογούμε διάφορα προγράμματα. και αν ήμασταν σίγουροι ότι υπάρχουν περισσότερες ανάγκες στην Ουγγάντα, φαντάζομαι ότι οι ίδιες ερωτήσεις μπορούν να θέσουν και άλλες ε, ε χώρες. Υπάρχουν πολλές ανάγκες. Το καταπιστευματικό ταμείο προβλέπει ε, έκτακτες, ε, δράσεις έκτακτες ανάγκες και το ζητούμενο είναι πώς μπορούμε να ε, αποσπάσουμε περισσότερη υποστήριξη, χρηματική υποστήριξη. Είναι δύσκολο για μας να πούμε πού ακριβώς διαδέθηκαν αυτά τα ποσά, γιατί στην Ουγγάντα το γραφείο του Πρωθυπουργού παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κρίσης και αυτή τη στιγμή ε, παρακολουθούν ε, την κατανομή των ε, χρημάτων. Νομίζω ότι αυτή την ερώτηση θα έπρεπε να την επευθύνατε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιούμαστε στον τομέα της αναψυχιακής βοήθειας και στο τομέα που αφορά το σύνδεσμο ανάμεσα στην ανθρωπιστική βοήθεια και την ανάπτυξη έχει δημοσιεύσει το Συμβούλιο ε, συμπεράσματα σχετικά. Η Ουγγάντα είναι πιλωτική χώρα και για την αναπτυξιακή συνεργασία και για το Σύνδεσμο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Ανάπτυξης. Τον Απρίλιο συμμετείχαμε σε ένα εργαστήριο στο οποίο συμμετείχαν τα κράτη-μέλη που δραστηριοποιούνται επί τόπου και από όπου και αν προέρχονται τα χρήματα, σημαντικό είναι να διατίθενται εκεί που είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες και να ε, καλύπτουμε τις ανάγκες των πιο ευάλωτων πληθυσμών, είτε είναι ντόπιοι πληθυσμοί είτε πρόσφυγες. Είναι Απαραίτητο λοιπόν να ε, μεταφέρουμε τα απαραίτητα ε, μηνύματα σε πολιτικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δύο άτομα από την ΕΚΟ. Ναι, πολύ σύντομα από την ανθρωπιστική άποψη δεσμευτήκαμε να δώσουμε 4,7 εκατομμύρια το 2017 έχουν διατεθεί όλα αυτά τα χρήματα τρέχουν τα προβλήματα ακόμα το 2018 ε, και ε, διαθέσαμε επιπλέον 24 εκατομμύρια. Οι κύριοι τομείς που καλύπτονται είναι αυτοί που αναφέρατε. Η εκπαίδευση, το υγιεινή, ε, η υγειονομική περίθαλψη, η ψυχολογική υποστήριξη που βρίσκονται στην καρδιά της ανθρωπιστικής δράσης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, να καλωσορίσω και τον Κλάου Στέρνς ε, που ήταν διευθυντής της ε, DG ECO. Ξέρω ότι στην Ουγκάντα έχετε πάει και τώρα σας βλέπω και σήμερα. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε όλους. Okay, we have one item left. Ένα θέμα έχουμε ακόμα που πρέπει να συζητήσουμε, είναι σημαντικό. Και ζητούμε από τους ερμηνείς ακόμη μερικά λεπτά. Okay, we move 18. Σημείο λοιπόν 18, ερώτηση της κυρίας Αρχεντίνη. Για τις δαπάνες που έχει η Επιτροπή δηλώσει ως ODA στην Επιτροπή Ντάκτουσα. Και μάλλον έχει κάπως ξαπνιαστεί και η Επιτροπή ΔΑΚ. Ποια είναι η κατάσταση. όλες οι δαπάνες προς την Τουρκία έχουν κοινοποιηθεί ως ODA. Δεν βλέπω ποιος είναι εδώ από την Επιτροπή και το όνομά σας παρακαλώ. Ζωγό Μλοχουά, από την ε, Ανάπτυξη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν έχουμε να κάνουμε με το καταπίστευμα για τους πρόσφυγες στην Τουρκία που θεσπίστηκε το 2016 κατόπιν των πολιτικών δεσμεύσεων που ανελήφθησαν με την δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία στο καταπίστευμα χρηματοδοτήτα απευθεία από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό με συμπληρωματικέ πρόσθετες συνεισφορέ από τα κράτη-μέλη τα οποία ε, οι οποίες συνεισφορμές ε, εισγράφονται στο καταπίστευμα ως ε, ειδικό εισόδημα. Καταγράφεται λοιπόν με την έκθεση του 2016 ως ODA το καταπίστευμα γιατί ο στόχος του είναι κατά κύριο λόγο είναι ανθρωπιστικός και περιβαλλοντικός με βάση τον ορισμό του ODA, δηλαδή επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Κατόπιν ε, αιτήματο κράτου μέλου, η γραμματεία DAC ζήτησε πρόσθετε πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανέλησε περισσότερο το καταπίστευμα σε λεπτομέρεια για να εξετάσει την αιρεσιμότητα. Η γραμματεία ήγηρε μια σειρά από ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον DAC συστήθηκαν σε λεπτομέρεια και στην ομάδα εργασίας για τις στατιστικές τον Ιανουάριο του 2018. Ε, τα συμπεράσματα κοινά για την ε, γραμματεία και όλα τα μέλη της Επιτροπής ΔΑΚ είναι τα εξής. Πρώτον, ότι είναι καταρχήν ε, επιλέξιμο ως ODA το σύνολο του καταπιστεύματος γιατί έτσι έχει οριστεί και με βάση και την οδηγία για την κοινοποίηση ΔΑΚ όπως αναφέρεται και όχι με βάση το γενικό πολιτικό, τη γενική πολιτική κατάσταση και όπως ορίζεται από, και, και επομένω το γεγονό ότι αυτό προβλέπεται στην ε, πολιτική συμφωνία και διακήρυξη με την Τουρκία δεν ορίζει το αν είναι ODA ή όχι. Επίσης 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του καταπιστεύματος του 2016 ε, έχουν αποκλείσει ε, δύο έργα ένα με τη Γενική Γραμματεία για τη διαχείριση μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας για την υποστήριξη της υποδοχής και ε, στήριξη των μεταναστών που επανέρχονται στη Τουρκία. Δεύτερον, μια άλλη, σύμβαση με τη Διεθνή Οργάνωση των Μεταναστεύσεων, IMO, IMO ε, σε σχέση με την ενίσχυση της τουρκικής ακτοφυλακής. Πρόκειται λοιπόν για συμβάσεις που απερίφθησαν, παρότι είχαν στόχους που θα μπορούσαν να προσαρμόζονται στη στόχευση, ωστόσο η γραμματεία ΝΤΑΚ θεώρησε ότι δεν ε, καλύπτουν τις προϋποθέσεις ODA, διότι ο πρωταρχικός στόχος είχε να κάνει περισσότερο με ευρωπαϊκές πολιτικές. Η γραμματεία ΝΤΑΚ λοιπόν όρισε μόνο ένα ποσοστό, 95% DAC, ODA ε, συγγνώμη, για όλα ε, στις πληρωμές του καταπιστεύματος του 2017. Δεύτερον, η αιρεσιμοεπιλεξιμότητα ODA θα ελέγχεται κάθε χρόνο από το 2017 και μετά, από τις χρηματικές ροές του 2017 και μετά. Φέτος το Μάρτιο η Γραμματεία ΝΤΑΚ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση για τις ροές 2017 του καταπιστεύματος, 36 συμβάσεις δηλαδή, 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και θεώρησε, εκτίμησε ότι ήταν κατά 100% επιλέξιμη ODA, ε, επιλέξιμες όλες οι ροές του 2017. Ενημερώθηκαν τα κράτη-μέλη για τα αποτελέσματα αυτά και... Μέχρι ε, τις παρούσες δεν έχει γίνει περαιτέρω συζήτηση επί I Ευχαριστούμε για την ε, απάντηση και συγχαρητήρια για το 97% υπαγωγή στην ΕΝΤΑΚ το 16 και πάνω ε, από, από αυτό το πόστο για το 17. Ναι, ναι, παρακαλώ όμως κάντε μας ένα χαρτί να μας στείλετε Έχουμε την συζήτηση του Ιανουαρίου των ε, Παρισίων από πρόκυψαν όλα αυτά. Ε, επίσης έχουμε ε, μία προφορική ερώτηση για την επόμενη ολομέλεια όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς πόρους που διατίθενται στην Τουρκία οπότε ίσως υπάρξει θέμα ή όχι για αυτή την δαπάνη του Οργανισμού Μετανάστευσης προς την συνοριοφυλακή. φυλακή. Εγώ υπέβαλα την ερώτηση γιατί ακριβώς ε, μου φαίνεται περίεργο και επίσης ανησυχώ. Έτσι το Κοινοβούλιο μπορεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να μάθουμε τι συμβαίνει. Να δούμε και στην Επιτροπή ΝΤΑΚ να δούμε τα κονδύλια πώς δαπανώνται. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να προχωρούμε και να έχουμε τέτοια τμηματική καταρρυπάς ενημέρωση με τις ερωτήσεις. Οπότε παρακαλώ όλα αυτά βάλτε τα σε ένα χαρτί να μας το διαβιβάσετε και να έχουμε επίσης ε, ε, συνημένα και τα υποστηρικτικά έγγραφα. Εμείς είμαστε η αρχή του προϋπολογισμού. Ήδη αρκετούς μπέλαδες έχουμε ε, για το για το θέμα του πώς δαπανώνται οι πόροι προβλέπονται στη συμφωνία με την Τουρκία. Η Επιτροπή ελπίζω ότι θα μας διαβεβαιώσει ότι θα στείλει αυτές τις πληροφορίες γιατί πρέπει να τις ζητήσουμε εγγράφος. Ναι, ναι, ναι. Σας τα διάβαζα από ένα έγγραφο και δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας ε, διαβιβάσω αυτό το που είχα τώρα. Όσον αφορά την ομάδα εργασία για αυτή την υποεπιτροπή της ΝΤΑΚ για τη στατιστική. Ε, συναντιέται αυτή η επιτροπή δύο-τρεις φορές ετησίως να δούμε τις ανάγκες και συνήθως η γραμματεία της ΝΤΑΚ έχει κάποιο είδου πρακτικά δεν είναι εμπιστευτική δεν είναι η κάμερα αυτή συνεδρίαση όπου το κοινοβούλιο μπορεί και αυτά τα πρακτικά να έχει διαθέσιμο. Ωραία, από το περιμένουμε αυτά τα εγγραφή και σας ευχαριστούμε. Και όπως η κυρία Σαρχιαντίνη, θέλουμε καλύτερη ενημέρωση για το τι γίνεται στην Πάμε τώρα στο 19, τα διάφορα. Δεν υπάρχει τίποτα από ό,τι ξέρω. Στο 20, επόμενη συνεδρίαση 25 Ιουνίου στις 3 η ώρα. Πέρα συνεδριά σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας συνάδελφοι και τους διερμηνείς.